God morgon och välkomna till vårt återupptagna utskottsmöte. Punkten 10 på dagordningen. Καλημέρα σας. Θα ήθελα να αρχίσουμε εμέσω. Το σημείο 10 είναι μια αναφορά σχετικά με την αποστολή στην Ισλανδία ε, από τις 29 μέχρι την 1η ε, Οκτωβρίου, 29 Σεπτεμβρίου μέχρι 1η Οκτωβρίου. Η κυρία Μπάουρ, η κυρία Σεμίσκη και η κυρία Κορνέλισαν μετέβησαν στην Ισλανδία. Και φυσικά ακολούθησαν και υπάλληλοι από την γραμματεία, από τις πολιτικές ομάδες αυτή την αποστολή. Θα ήθελα Εν συντομία να σας πω για ποιο λόγο διοργανώθηκε η αποστολή. Θέλαμε να αποκτήσουμε ε, περισσότερες γνώσεις σχετικά με την νομοθεσία και την πρωτοβουλία που αναλύθηκε στην Ισλανδία σχετικά με τα θέματα ισότητας των φύλων. Έγιναν πολλές συζητήσεις σε προηγούμενες συνεδριάσεις που κάναμε για την άδεια μητρότητας, ε, πατρότητας και τη γονική άδεια. Εφόσον ήταν εξαιρετικά επίκαιρο το θέμα, φυσικά και για την Επιτροπή μας. Φυσικά ενημερωθήκαμε για την οικονομική κρίση που έπληξε σφόδρα την Ισλανδία. Επίσης ε, μάθαμε ότι υπάρχει μια ειδική επιτροπή που ασχολείται ακριβώς με αυτό το θέμα, να εξετάσει δηλαδή τις συνέπειες της κρίσης, με ποιο τρόπο επηρεάζονται οι γυναίκες και οι άντρες από την κρίση. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η αποστολή. Έχουμε εκδώσει και ένα ανακοινωθέν τύπου επ' αυτού και μετά την αποστολή είναι διαθέσιμο και επίσης ε, στις, ε, στους φακέλους σας ε, υπάρχει και ένας κατάλογος των συνεδριάσεων που είχαμε επί τόπου. Εν συντομία θα ήθελα να σας πω κάποια πράγματα για τις διάφορες συνεδριάσεις που κάναμε. Συναντηθήκαμε με τον ε, Υπουργό ε, Υγείας ε, και Κοινωνικών Υποθέσεων και Απασχόλησης της Ισλανδίας και άλλα κυβερνητικά στελέχη. Η αποστολή μας συνέπεσε με την παρουσίαση από πλευράς της κυβέρνησης του σχεδίου προϋπολογισμού. Ε, και ήταν πολύ θυελώδης ε, οι συζητήσεις λόγω των δημοσιονομικών περικοπών, λόγω φυσικά της ε, χρηματοπιστωτικής κρίσης. Πάντως ήταν θετικό το ότι όλοι οι υπουργοί της κυβέρνησης μέσα στον προϋπολογισμό έχουν ειδικά σχέδια για την ισότητα των δύο φύλων για το 2011. Επίση, ενημερωθήκαμε την κυβέρνηση γενικότερα για την κατάσταση στην Ισλανδία, εστιάζοντα φυσικά στα θέματα που μα ενδιαφέρουν, δηλαδή ε, την ισότητα των δύο φύλων. Ένα θέμα που συνιστά προτεραιότητα, τονίζω, για την Ισλανδική κυβέρνηση. Ε, προετοίμασαν το πέμπτο σχέδιο δράση ε, για την ισότητα των φύλων. Επίση, μάθαμε πω ε, για αυτό το θέμα τη ισότητα στην Ισλανδία υπάρχει, υπάρχουν πάρα πολλά πολλά στελέχη κυβερνητικά που ασχολούνται με αυτό το θέμα, τέσσερις υπουργοί συγκεκριμένα ε, για τις κοινωνικές υποθέσεις, ε, για τη δικαιοσύνη, για τα οικονομικά και ο Πρωθυπουργό ε, έχουν επιληφθεί του ζητήματος σε υψηλό επίπεδο λοιπόν ασχολούνται με το θέμα της ισότητας των δύο φύλων. Επίσης επισκεφτήκαμε τη Βουλή της Ισλανδίας, συναντηθήκαμε με τον πρόεδρο της Επιτροπής αρμόδιας για τα θέματα ισότητας και πολλά, πολλοί βουλευτές του, της Βουλής της Ισλανδίας συμμετέχουν σε αυτήν την ειδική επιτροπή και ήταν παρόντες και ως εκ τούτου ενημερωθήκαμε διεξοδικά για το θέμα της ισότητας των δύο φύλων. Επίσης συναντηθήκαμε με το Ινστιτούτο Ισότητας των Δύο Φύλων της Ισλανδίας και ενημερωθήκαμε για τις εργασίες του Ινστιτούτου. Αυτή η παρουσίαση επίσης υπάρχει ε, στην ιστοσελίδα της Επιτροπής μας και μπορείτε να ενημερωθείτε. Επίσης συναντηθήκαμε με εκπροσώπους κοινωνίας των πολιτών και διαφόρων και να σας πω επίσης ότι ε, συναντήκαμε τον πρόεδρο και ιδρυτή ε, μιας χρηματοπιστωτικής εταιρείας, ε, μιας χρηματοπιστωτικής εταιρείας που ιδρύθηκε για να υπάρχει μια γυναικεία άποψη για αυτό το κομμάτι της οικονομίας, να εξετάζουμε αυτό το κομμάτι της οικονομίας από, μέσα από ένα γυναικείο πρίσμα και μας εξήγησαν ε, τις δράσεις ε, αυτού του Ινστιτούτου, αυτή, αυτές της εταιρείας που λέγεται Auro Capital και απεδείχθη ότι αυτή η εταιρεία είναι ιδιαίτερα επιτυχής ε, ως προς τα χρηματοπιστωτικά ε, ήταν πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον, διότι διαπιστώσαμε ότι είναι δυνατόν να υπάρχουν τέτοιες χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες, αλλά να συνδυάζονται με μία ε, να συνδυάζεται δηλαδή αυτή η καλή επιχειρηματική δραστηριότητα μαζί με το σεβασμό των αρχών της ισότητας των δύο φύλων. Επίσης, μια άλλη οργάνωση, η που ασχολείται με την εκπαίδευση, την παροχή συμβουλών προς αυτούς που έχουν βιώσει σεξουαλική βία, σεξουαλικές επιθέσεις. Συναθήκαμε μαζί τους και παρότι έχει τόσο μεγάλη βερίτα το θέμα της ισότητας των δύο φύλων, όπως απεδείχθη από όλη τη συνεργασία που είχαμε με την Ισλανδική κυβέρνηση, παρόλα αυτά εξακολουθούν να υπάρχουν πελώρια προβλήματα ε, ως προς τη βία κατά των γυναικών. Έτσι μάθαμε επίσης, ε, ε με μια οργάνωση που λέγεται Skotrum και είναι μια ε, πολύ γνωστή οργάνωση μεταξύ άλλων διότι κάθε χρόνο αναλαμβάνει πρωτοβουλίες στα τέλη Οκτωβρίου ε, και διοργανώνει διαδηλώσεις ε, για ε, τους ίσους μισθούς, για τις γυναίκες και οι γυναίκες πάβουν την εργασία τους τότε, δηλαδή απεργούν εκείνη την ημέρα για να ε, δείξουν ότι ε, λαμβάνουν χαμηλότερες αμοιβέ ε, σε σχέση με τους άντρες και βλέπουμε λοιπόν ότι έχουν γίνει σοβαρές προσπάθειες στην Ισλανδία για να καταπολεμηθεί αυτό το πρόβλημα τα τελευταία 13 χρόνια. Επίσης συναντηθήκαμε με τους ε, αρμόδιους για τις διαπραγματεύσεις της Ισλανδίας για την προσχώρηση της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, αυτά είναι συντομία ήταν πραγματικά εξαιρετικά αξιόλογη αυτή η αποστολή και τώρα θα ήθελα να σας δώσω τη δυνατότητα αν θέλετε να κάνετε ερωτήσεις ή κάποια σχόλια σχετικά με την αποστολή της Αντιπροσωπής Επιτροπής ε, των Γυναικών. Η κυρία Μπιλμπάου έχει ζητήσει το λόγο, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Μόνο μία ερώτηση θα είχα για μία έκθεση που διάβασα πριν από κάποια χρόνια. Η αντίφαση σε σχέση με τις βόρειες χώρες όσον αφορά τα πιο προηγμένα μέτρα υπέρ της ισότητας ακόμα και τις προτάσεις που είναι τόσο ενδιαφέρουσες και ακούσαμε και εφαρμόζονται. Όμως ωστόσο η ανάπτυξη αυτού του προγράμματος για την ισότητα βρίσκεται σε αντίφαση με τους υψηλούς δείκτες βίας που υπάρχει, υπάρχουν σε αυτή τη χώρα. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω πώς γίνεται αυτό έχετε την ευκαιρία, είχατε την ευκαιρία να μάθετε και να γνωρίσετε τα ποσοστά της βίας κατά των γυναικών στη χώρα αυτή και αν έχουν αντιμετωπιστεί και έχουν διαπιστωθεί τα πραγματικά αίτια. Διότι υπάρχει μια τόσο ανεπτυγμένη κατάσταση όπως αυτή στις βόρειες χώρες για την ισότητα. Από την άλλη όμως πλευρά η αύξηση ή ο αριθμός που είναι τόσο υψηλός των περιπτώσεων βίας κατά των γυναικών. Ε, Κυρία Παπαδοπούλη, παρακαλώ. Φαίνεται ότι ήταν αρκετά ενδιαφέρουσα η επίσκεψή σα στην Ισλανδία. Πριν από μερικά χρόνια είχαμε επισκεφθεί αυτή τη χώρα ω Επιτροπή Γυναικών του Συμβουλίου τη Ευρώπη, γιατί πραγματικά τα σχέδια που έχουν για την πατρογονική άδεια, τη μητρική άδεια, την άδεια πληρώνονται. Και αυτό ήταν κάτι εντυπωσιακό γιατί σε σύγκριση με άλλε ευρωπαϊκέ χώρε, η Ισλανδία ήταν η μόνη χώρα που επλήρωνε τον πατέρα για να μείνει στο σπίτι με πατρογονική άδεια. Διερωτούμε πώς η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει ε, αυτό συγκεκριμένα το θέμα. Αν έχουν αλλάξει πολιτική, αν εξακολουθούν να πληρώνουν τον πατέρα για να μείνει στο σπίτι όταν τεκνοποιεί η σύζυγος, πώ ε, πώς έχει επηρεάσει η οικονομική κρίση αυτόν ακριβώς το ρόλο του πατέρα να πληρώνεται κιόλας για να μείνει στο σπίτι. Ευχαριστώ. θα προσπαθήσω εν συντομία να σα απαντήσω σε αυτά τα ενδιαφέροντα ερωτήματα. Κυρία Μπιλμπάου, για τι βαθύτερε αιτίε σχετικά με τα τα αυξημένα, εξαιρετικά αυξημένα επίπεδα βίας σε, αυτά, σε αυτές τις χώρες, παρότι είναι σχετικά ε, ικανοποιητική η νομοθεσία για τα θέματα ισότητας των φύλων. Λοιπόν, για την Ισλανδία δεν ε, καταφέραμε να ε, αποκτήσουμε έτσι συγκεκριμένες πληροφορίες που θα εξηγούσαν γιατί εξακολουθούν να υπάρχουν τόσα πολλά περιστατικά βίας στην Ισλανδία. Ε, Επίση, κάτι που συζητήσαμε, δεν ξέρω αν είναι η βασική αιτία, αλλά είναι μία αιτία, τέλο πάντων αναφέρθηκε στι συζητήσει μα. Ε, πρόκειται λοιπόν για τη συνειδητοποίηση ότι καταγγέλλεται ε, η βία κατά των γυναικών λόγω αυτής της νομοθεσίας που υπάρχει και επειδή υπάρχει δυνατότητα καταγγελίας αυξάνεται ο αριθμός των καταγγελιών. Ταυτόχρονα ε, μπορεί να σκεφτεί κανείς ότι ναι, είναι ικανοποιητική νομοθεσία και ως εκ τούτου δηλαδή αυξάνει τη συχνότητα των καταγγελιών μέσα ε, στα τατιστικά στοιχεία ε, προκύπτουν κάποιες τέτοιες ενδείξεις, ε, μπορεί να αποτελεί αυτό μία από τις αιτίε, αλλά δεν ε, μάθαμε ε, πάρα πολλά πράγματα για τις υπόλοιπες βασικές αιτίε του φαινομένου. Κυρία Παπαδοπούλου, για την οικονομική κρίση και πώς επηρέασε αυτό την δυνατότητα που υπάρχει για την γονική άδεια, άδεια μητρότητας μάθαμε λοιπόν ότι λόγω της κατάστασης ε, της δημοσιονομικής, λόγω της κρίσης, η κυβέρνηση πρότεινε στο σχέδιο προϋπολογισμού για το 2011 να διατηρήσει την άδεια για του, την άδεια πατρότητας ε, αλλά λόγω της ε, ε, τωρινής κατάστασης υπήρχε και μία πρόταση να μειωθεί ο αριθμός των μηνών για την γονική άδεια συνολικά. Σας υπονθυμίζω ότι είχαν προταθεί ε, οι δύο μήνες, δηλαδή να μειωθεί κατά δύο μήνες η γενικότερα η γονική άδεια. Αλλά πάντως ε, η άδεια πατρότητας ε, διατηρείται μέσα στο σχέδιο προϋπολογισμού. Αν δεν υπάρχουν τώρα άλλες ερωτήσεις, σας προτείνω να περάσουμε στο επόμενο σημείο της ε, ημερησίας διατάξεως, ε, ε, δηλαδή στην ψηφοφορία για διάφορες εκθέσεις. Η πρώτη φέρει επί της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενσωμάτωση των Ρωμά. Στη χτεσνή μας συνεδρίαση κάναμε τη συζήτηση για αυτό το θέμα. Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών είναι η καθήλυνα αρμόδια. Η συγγήτρια, η κυρία για ΡΟΚΑ πρότεινε να εγκρίνουμε τις τροπολογίες εδώ στη δική μας Επιτροπή, ώστε να υποβληθούν στη συνέχεια στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών. Θα σας δώσω το λόγο ε, πριν αρχίσουμε την ψηφοφορία. Παρακαλώ. Thank you very much, Madam Chair. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Χθε συζητήσαμε αυτό και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις προτάσεις σας Είχα μια πολύ καλή πρόταση από την κυρία σε ενός πρόταση για την ανταλλαγή των πρακτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και έτσι με αυτό το πλαίσιο μπορώ να πω γενικεύω την έκθεσή μου και την εξειδικεύω και σε σχέση με τα σημεία για το, τον κατάλογο ψηφοφορίας όσον αφορά τις ε, τροπολογίες ε, κατά τη συζήτηση που είχαμε χθε έχουν γίνει αυτές οι αλλαγές και θα ήθελα να σας ζητήσω αυτό το κείμενο να είναι πολύ πιο στοχοθετημένο όσον αφορά τη διάσταση του φύλου. Όσον αφορά για τη στρατηγική της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους τσιγκάνους, πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι στόχοι αυτής της στρατηγικής θα συνδέονται σε υψηλό βαθμό με τους στόχους ε, του έργου της δικής μας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. Και ως εισηγήτρια θα κάνω ότι περνάει από το χέρι μου και ζητώ τη συνεργασία για τα επόμενα χρόνια. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Γιαρόκα. Μπορούμε ομαδών να ψηφίσουμε για όλες αυτές τις ε, τροπολογίες. Ε, υπάρχουν αντιρρήσεις. Ε, μπορούμε να ψηφίσουμε τις τροπολογίες ομαδών. Όχι, δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. Πολύ ωραία. Τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά... Ένα και δύο. Αυτή είναι η αριθμή των τροπολογιών, τι οποίε θα ψηφίσουμε από κοινού. Με ανάταση χειρό, παρακαλώ, ψηφίστε υπέρ. Κατά τώρα. Αποχές εγκρίνονται. Σας ευχαριστούμε, κυρία Γιαρόκα. nästa ärende är eh, genomförande av ett fördjupat samarbete. Τώρα, ε, θέσπιση ενισχυμένη συνεργασία στον τομέα του δικαίου που είναι εφαρμοστέ στο διαζύγιο και τον δικαστικό χωρισμό. Ε, η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων, η καθήλια αρμόδια επιτροπή, Ε, ξεκίνησε αυτό το θέμα από 14 κράτη-μέλη και κατόπιν προσχώρησαν στην ενισχυμένη συνεργασία και άλλα κράτη-μέλη. Ο στόχος είναι να διευκολύνουμε ε, όσους έχουν συνάψει γάμους με ανθρώπους ε, άλλης υπηκότητας και δίνουμε τη δυνατότητα μεταξύ άλλων στους συντρόφους να επιλέξουν το εφαρμοστέο δίκαιο και φυσικά και οι ε, δύο σύζυγοι ενημερώνονται για, την, ε, ε, για το εφαρμοστέο δίκαιο, την εφαρμοστέα νομοθεσία. Η κυρία Νίμπλερ είναι η συντάκτρια, αλλά δυστυχώς ε, είναι σε ένα αεροδρόμιο στο Μόναχο, αν δεν κάνω λάθος, η κυρία Νίμπλερ ε, και δεν μπορεί να πετάξει λόγω της ε, χιονόπτωσης. Έχει αποκλειστεί λοιπόν στο Μόναχο και δεν μπορεί να είναι μαζί μας σήμερα για να κάνει κάποιες παρατηρήσεις για το θέμα αυτό. Ε, την ενημερώσαμε πάντως και μας είπε ότι παρόλα αυτά μπορούμε να ψηφίσουμε σήμερα. Αν δεν υπάρχουν ερωτήσεις, σας προτείνω ευθύ αμέσω ε, να περάσουμε ε, στην ψηφοφορία για την πρόταση τροποποιημένης νομοθεσίας για τα διαζύγια και τους δικαστικούς χωρισμούς. Δεν βλέπω να υπάρχουν αντιρρήσεις. Ας αρχίσουμε λοιπόν. Τροπολογία 4 υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται 5 υπέρ ε, κατά αποχές εγκρίνεται η 14 καταπίπτει οπότε 15 υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία υπαριθμών 1 υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, οι 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 9 καταπίπτει. Ε, ψηφίζουμε για την 10 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, έλεγχος παρακαλώ, ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίστε παρακαλώ. Για την 10. Ψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. ισοψηφία 11 προς 11, άρα απορρίπτεται. Η 11 τώρα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 12 έχει αποσυρθεί. 3 υπέρ παρακαλώ, κατά αποχές εγκρίνεται και 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και η τελική ψηφοφορία του σχεδίου γνωμοδότησης ψηφίστε παρακαλώ ψήφισαν όλοι πέρας εγκρίνεται με 20 ψήφους υπέρ και δύο αποχές Συγχαρητήρια κυρία Νίμπλερ που είσαστε στο Μόναχο αποκλεισμένοι. Och vi har ju beslutat om ändringar på ε, χτες θυμάστε είχαμε αποφασίσει να κάνουμε κάποιες αλλαγές στη μερίσια διάταξη οπότε ε, έχουμε αφαιρέσει το σημείο 13 και τα σημεία 14 και 15 αναβλήθηκαν για την επόμενη συνεδρίαση γι' αυτό το λόγο περνάμε στο σημείο 16 Πρόκειται για τη μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η καθήλυνα αρμόδια επιτροπή είναι η Επιτροπή Περιβάλλοντος όπου η κυρία Εστρέλα είναι η εισηγήτρια. Η δική μας εισηγήτρια είναι η κυρία Γκυγιόμ. Ε, ο στόχος της γνωμοδότησής μας είναι να τονίσουμε όλος ιδιαιτέρως τις ανισότητες στον τομέα της υγείας, κυρίως ως προς την γυναική υγεία θα ήθελα πριν ε, προβούμε στην ψηφοφορία να δώσω το λόγο στην κυρία Γκυγιόμ. Παρακαλώ. Δεν είναι εδώ η κυρία Γκυγιόμ. Η κυρία πείτε και να έχει ζητήσει το λόγο. Thank ε, Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για την πολύ καλή έκθεση και να κάνω μια αποσαφήνιση σε σχέση με το ΕΡΚ στις τροπολογίες 52 και 83 σε τμήματα ψηφοφόρια ε, ζητήθηκε όπου η θέση του ΕΡΚ είναι να καταψηφιστεί η άμβλωση, οι εκτρώσεις να καταψηφίζουν εγώ θα είμαι υπέρ και των δύο τροπολογιών προσωπικά και για το θέμα της πρόσβασης σε ε, ε δυνατότητες ε, να χρησιμοποιούνται ε, φυλακτικά και για τις τροπολογίες 84, 88, 96, 98, 90, 20, 21 ελεύθερη ψήφος από πλευράς του ΕΛΚΑ προσωπικά εγώ θα υπερψηφίσω αυτές. Ευχαριστώ για την κατανόηση και για την δυνατότητα να αποσαφινιστούν αυτές οι διαφορετικές, οι ε, διαφοροποιημένες θέσεις σε αυτά τα θέματα. Μάλιστα σας ευχαριστούμε. Η κυρία Εστρέλα έχει τώρα το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Εμείς συζητήσαμε χτες το σχέδιο έκθεσης στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Ήταν μια συζήτηση που συμμετείχαν σε αυτήν πάρα πολλοί ευρωβουλευτές και ήταν πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Έγιναν προτάσεις όπως διατυπώθηκαν από τους συναδέλφους που συμμετείχαν στη συζήτηση, προτάσεις που θα εμπλουτίσουν τη δική μου πρόταση, τη σχέδιο έκθεσης. Η προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών <clears throat> λίγη στις 10 του μήνα σε σχέση με τη γνωμοδότηση της κυρίας Γκυγιώμα, είναι μια γνωμοδότηση που θεωρώ ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα και επαρκής κιόλας ε, όσον αφορά την προοπτική της Επιτροπής ε, Δικαιωμάτων Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Μια και επικεντρώνεται στις ε, πιο σημαντικές ανισότητες όσον αφορά την υγεία υπό το πρίσμα του φύλου, υπό το πρίσμα των γυναικών. Και είχαμε και αυτή τη συζήτηση και εδώ και εξάλλου από πλευρά του Ζορβάν που είναι ε, σκιώδης εισηγητής ε, όσον αφορά την Επιτροπή Περιβάλλοντος ε, και η ιατρός έχει μια προοπτική θα έλεγα πολύ σημαντική στις απόψεις του και που συμπληρώνει σίγουρα τις άλλες προοπτικές και προτάσεις ώστε μπορούμε να πούμε ότι εμείς είμαστε σε θέση να ταυτοποιήσουμε και να εντοπίσουμε με αυτόν τον τρόπο ποιες είναι οι ανισότητες που εξακολουθούν και υφίστανται όσον αφορά τις διαφορές ε, μεταξύ ανδρών και γυναικών στην αντιμετώπιση, στην πρόσβαση, στην περίθαλψη και στις υπηρεσίες υγείας. Και όλα αποκαλύπτουν ότι η ίδια η μακροζωία είναι διαφορετικές για το προσδόκιμο ζωής. Έχουν μεγαλύτερη ζωή, μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής οι γυναίκες και υπάρχει μεγάλη διακύμανση όσον αφορά την κατάσταση στα κράτη-μέλη. Επίσης αναφερθήκαμε, αναφέρθηκε ότι τα φάρμακα δεν έχουν τις ίδιες επιπτώσεις ακριβώς στις γυναίκες και τους άνδρες και τα λοιπά. Είναι μια συζήτηση λοιπόν πολύ ενδιαφέρουσα αυτή. Θα ήθελα να κάνω μια έκκληση σε σχέση με αυτό που αναφέρθηκε από την προλαλή σας πιο πριν και να πω ότι η Επιτροπή ψηφίζει αυτές τις σχέσεις όσον αφορά την αναπαραγωγική υγεία και αυτή είναι μια διαφορά πάλι σε σχέση με τη βιολογική διαφορά και ανατομική διαφορά και την φυσιολογική διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών, σωματικές διαφορές και άλλες, βιολογικές και άλλες. Αυτές οι διαφορές λοιπόν θα πρέπει να αναγνωριστούν και να γίνουν αποδεκτές από την Επιτροπή. Απευθύνω έκκληση λοιπόν να τις υπερψηφίσουμε αυτές τις προτάσεις, αυτές τις τροπολογίες που αφορούν ακριβώς την υγεία, την σεξουαλική υγεία, την αναπαραγωγική υγεία των γυναικών. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κυρία Εστρέλα. Κυρία Γκυγιόμ, ε, ζητώ συγγνώμη που κατέφθασα αργοπορημένη, αλλά είμαι μέλος σε τρεις επιτροπές και συνεδριάζουν ταυτόχρονα. Έτσι, την ίδια ώρα, την ίδια ημέρα. Ε, ψήφιζα τώρα για την ε, πρωτοβουλία των πολιτών. Νομίζω ότι είναι επίσης σημαντικό θέμα. Ζητώ συγγνώμη, ξέχασα και την ηλεκτρονική μου κάρτα παρεπιπτόντος από το τρέξιμο. Θα ήθελα ε, για αυτή την έκθεση που ψηφίζουμε σήμερα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν ευρύτατα για την ε, σύνταξη των τροπολογιών. Υπήρχε σχετικά μεγάλη ομοθυμία και αυτό καταδεικνύει το ενδιαφέρον που παρουσιάζει αυτό το θέμα της υγείας των γυναικών, κυρίως τη μείωση των ανισοτήτων. Ε, και προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε ένα τον άλλον ως προς τις απόψεις μας. Ε, μπορέσαμε για την πλειοψηφία δε των ε, επιμέρους σημείων της έκθεσης να καταλήξουμε σε κάποιους συμβιβασμούς. Ελπίζω να έχει έσει έκβαση η ψηφοφορία για την γνωμοδότηση αυτή που θα ενταχθεί στην βασική έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Πρόεδρος, ευχαριστούμε κυρία Γκυγιώμη. Η κυρία Λούλινγκ τώρα. Μάλιστα, πρόεδρε, ευχαριστώ. Εγώ μόλις είδα τις συμβαστικές ε, τροπολογίες και θα ήθελα να αναφερθώ στην πρώτη συμβαστική τροπολογία Έχω επίγνωση του ότι πρέπει να καταλήξουμε συμβαστικές τροπολογίες και να συμπεριλάβουμε τις απόψεις όλων στο μέτρο του δυνατού, αλλά ε, δεν είναι εύληπτη. Αυτή η πρώτη συμβαστική τροπολογία όπως έχει συνταχθεί δεν νομίζω να μπορούμε να, να υποβάλουμε μια τέτοια τροπολογία. Δεν θα καταλάβει κανείς. Επίσης, ε, συμβαστική τροπολογία 6. Λέει εδώ και διαβάζω στα αγγλικά ε, ότι τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κατοχυρώσουν τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία των γυναικών και να λάβουν υπόψη ε, την θνησιμότητα των γυναικών στις πολιτικές τους και να παράσχουν τη δυνατότητα ασφαλούς άμβλωσης εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι πηγιώνται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πώς θα το επιβάλλετε αυτό. Δεν είναι, δεν άπτεται των αρμοδιοτήτων μας. Σας ευχαριστούμε κυρία Λούλινγκ. Η ε, κυρία Γκαρσία Πέρες τώρα. Εγώ πιστεύω ότι έχοντας συνειδητοποιήσει το δικό μας επίπεδο αρμοδιοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούμε να θεσπίσουμε, να συγκροτήσουμε τα δικά μας υγειονομικά συστήματα όπου θα διασφαλίζουμε την υγειονομική ασφάλεια τα, στα θέματα μ, αναπαραγωγής, αναπαραγωγικά θέματα και σεξουαλικής υγείας αλλά και σε συνεργασία με άλλα κράτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε φυσικά τα θέματα που αφορούν τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία είναι θεμελιώδους σημασίας. Υπάρχουν εκατομμύρια γυναίκες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που καθημερινά βρίσκονται σε κίνδυνο κινδυνεύει η ζωή τους και η υγεία τους επειδή δεν έχουν πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες που να διασφαλίζουν αυτή την υγεία όπως πρέπει και γι' αυτό επίσης στο μέτρο που η δική μας πολιτική συνεργασίας μπορεί να προχωρήσει σε αυτό το επίπεδο πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα γίνεται αυτό σε σχέση με άλλε χώρες. Υπάρχουν παραδείγματα για προγράμματα που δρομολογούνται με τα ευρωπαϊκά κονδύλια και τα ευρωπαϊκά προγράμματα με αυτέ τι χώρες με ιατρικέ οργανώσει, οργανισμού υπέρ των γυναικών και έτσι υπάρχει ε, σε αυτό το επίπεδο συνεργασία. Ευχαριστούμε κύριε Πίτικενεν. To... Θα ήθελα να αναφέρω ένα ε, σημείο διευκρινιστικό. Στους στόχους της χιλιετίας ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύτηκε Και βεβαίω ο στόχος που δεν έχει εκπληρωθεί καθόλου είναι η υγεία των ε, μητέρων ε, και η αναπαραγωγική υγεία ε, στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό, αυτός ο στόχος πρέπει να επιδιωχθεί μέσα από διάφορε μεθόδους συνεργασίας. Η κυρία Τόμψεν. Και εγώ θα ήθελα να προσθέσω ότι και εμείς συμμετέχουμε στην στρατηγική των ΗΕ με στόχο την Ε, θα θέλαμε και εμείς να συμβάλλουμε στην περιορισμού της θνησιμότητας μητέρων ε, σαν στόχο. Σα uh, um, Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Λούλινγκ ε, έθεσε ένα ερώτημα. Πώς μπορεί κανείς να επιβάλλει κάτι τέτοιο εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. η συνθήκη της Λισαβόνας λέει ότι δεν θα πρέπει να επηρεαστεί το θέμα της άμβλωσης κάνετε, δίνετε διάφορες υποσχέσεις και εάν επανέλθετε σε αυτές τις υποσχέσεις τότε η συνθήκη της Λισαβόνας θα πρέπει να εγκαταλείψει την ίδια τη συνθήκη γιατί με τον τρόπο που πέρασε η συνθήκη της Λισαβόνας ήταν ότι έγιναν υποσχέσει ότι δεν θα υπάρξει καμία νομοθεσία επί του θέματο Η κυρία και η κυρία Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα κι εγώ να θίξω για άλλη μια φορά ένα θέμα το οποίο είναι η συμβαστική πρόταση υπαριθμών 6 που συζητήθηκε εδώ. Η ομάδα του ΕΛΚ ζήτησε ψήφους κατά τμήματα στο σύνολο αυτής της πρότασης. Στο πρώτο τμήμα να έχουμε ελεύθερη ψήφο και κατόπιν να εκπροσωπηθεί η επίσημη θέση Γι' αυτό λοιπόν επιθυμώ να επαναφέρω το θέμα αυτό, ή δυνατόν. Όσον αφορά δηλαδή αυτή τη συμβαστική πρόταση, να ψηφίσουμε κατά τμήματα. Θα ήθελα η πρόταση αυτή να αναφερθεί ε, στον ε, πρόεδρο και στους συναδέλφους. Και αυτό το θέμα, αυτή την πρόταση την υποβάλλω εκ μέρους της πολιτικής μας ομάδας για να τη λάβετε υπόψη σας. Ευχαριστώ και πριν δώσω το λόγο στην κυρία Λούλινγκ θα ήθελα να διευκρινίσω κάτι. Βάσει του κανόνα 160 ε, του ιστορικού κανονισμού για τις αρχές που διέπουν τις ψηφοφορίες δεν είναι δυνατόν να κάνουμε τμήματική, κατά τμήματα ψηφοφορία όταν ψηφίζουμε για μια συμβαστική τροπολογία. Αυτό δυνάμει το ιστορικού κανονισμού. Ήθελα να σας ενημερώσω για να είναι σαφές. Κυρία Λούλινγκ, παρακαλώ. Πρόεδρε, εγώ καταλαβαίνω ότι στα πλαίσια της αναπτυξιακής μας πολιτικής θα έπρεπε να παρακινήσουμε να ενθαρρύνουμε οι χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δρουν κατά αυτόν τον τρόπο. Αλλά τι λέει μέσα στο συμβαστικό κείμενο στα αγγλικά έτσι και το τα καταλαβαίνω λίγο τα αγγλικά. Λέει, η Ευρωπαϊκή τα κράτη-μέλη θα πρέπει να παράσχουν τη δυνατότητα ασφαλούς άμβλωσης μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό εντάξει, μπορούν να το κάνουν. Και beyond, λέει, και πέραν της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορούμε εμείς να παράσχουμε τέτοια δυνατότητα εκτός. Δεν έχουμε τέτοια αρμοδιότητα. Μπορούμε να τους ενθαρρύνουμε να εφαρμόσουν παρεμφερή πολιτική, αλλά δεν μπορούμε, τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να ε, δώσουν αυτή τη δυνατότητα δεν μπορούμε να καταψηφίσουμε, αλλά αν θέλετε να το πράξουμε... Και διακόπτει κυρία Λούλη. Ναι, τώρα φτάσαμε στη στιγμή της ε, ψηφοφορίας, αλλά πρώτα ε, θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Σεμάνσκι. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν νομίζω ότι θα έπρεπε να παρασυρθούμε από συναισθηματική φόρτιση εδώ από συναισθήματα. Υπάρχει μια λογική εδώ και υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο και ένα γεωγραφικό πλαίσιο. Δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτά τα πλαίσια. Έτσι. Αυτό για το οποίο συζητάμε είναι ο κόσμος στο σύνολό του παγκόσμια. Συμφωνώ λοιπόν με την κυρία Λούλινγκ σε αυτά που είπε τα κράτη-μέλη πραγματικά υποτίθεται και πρέπει να επιβάλλουν αυτά εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν γίνεται αυτό και έχουμε και τους συμβιβασμούς. Συμβιβασμοί, συμβαστικές τροπολογίες είναι προσπάθεια να εξευρεθεί μια διατύπωση που η συντριπτική πλειοψηφία θα μπορεί να δεχθεί. Μου φαίνεται ότι αυτή η διατύπωση λοιπόν δεν είναι συμβιβαστική διατύπωση που μπορεί να υποστηρίξουν όλοι. Το ΕΛΚ δεν θα υποστηρίξει, δεν θα υπερψηφίσει αυτό το αίτημα. Είναι μια διατύπωση που είναι μια συγκρουσιακή θα έλεγα διατύπωση για ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, το θέμα της υγείας. Στην δική μου τη χώρα, την Πολωνία, ο νόμος είναι σαφέστατος και κάθετος για τις αμβλώσεις. Το ίδιο το συνταγματικό δικαστήριο γνωμοδότησε σχετικά για αυτό το θέμα και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να σέβεται το γεγονός ότι οι συγκεκριμένες χώρες, κάποιες χώρες όταν προσυπέγραψαν και ενέκριναν τη συνθήκη της Λισαβόνας διατήρησαν κάποιες επιφυλάξεις ως όρους και προϋποθέσεις και επέμειναν, ενέμειναν ο δικό, η δική τους νομοθεσία να πριτανεύσει και να είναι σεβαστή. Νομικές τώρα διατάξεις που θα απαιτούν από τα κράτη-μέλη να δράσουν ενάντια σε αυτό το νομοθετικό πλαίσιο δεν συνάδουν ούτε με την, την ανεκτικότητα ούτε με πνεύμα συμβιβασμού. Οπότε Γι' αυτό λοιπόν θα έλεγα σέβομαι άλλε απόψεις, ε, διαφορετικές απόψεις. Σε αυτή την περίπτωση όμως έχουμε συγκρουσιακή σύγκρουση συμφερόντων. Πριν δώσω το λόγο στην Εστρίλα που είναι η τελευταία ομιλήτρια, ε, θα ήθελα να σας πω ότι θα ψηφίσουμε για την ε, συμβαστική τροπολογία Τέλο πάντων, θα περάσουμε τώρα ευθύ αμέσω στην ψηφοφορία, αλλά θα δώσω το λόγο στην κυρία Εστρέλα, γιατί είναι αρμόδια για το θέμα στην Επιτροπή περιβάλλοντο. Παρακαλώ. Σα ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό να αποσαφηνίσουμε κάποια σημεία. Αυτό το οποίο εμπεριέχεται σε αυτό το συμβιβασμό υπαριθμών 6 ήδη εγκρίθηκε σε άλλα έγγραφα, με άλλα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τώρα προφανώς δεν, δεν είναι υποχρεωτικό τα κράτη-μέλη να τροποποιήσουν την δική τους αντίστοιχη νομοθεσία. Καθόλου. Μία σύσταση υπάρχει μόνο για τα κράτη-μέλη. Σύσταση. Και υπενθυμίζω εδώ ότι επανειλημμένα κατά τη διάρκεια αυτών των τελευταίων ετών <clears throat> εγκρίθηκαν ταυτόσιμες παρόμοιες συστάσεις από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εντάξει. Δεύτερο τώρα. Κατά δεύτερο λόγο <clears throat> υπάρχουν ευθύνε ε, όσον αφορά τρίτες χώρες. Όχι μόνο για την υποστήριξη που οφείλουμε να δώσουμε για την ανάπτυξη στις χώρες αυτές, αλλά και επειδή συμμετέχουν με τη συμμετοχή στους ορισμούς και προσανατολισμούς των Ηνωμένων Εθνών, είμαστε μέρος εμείς αυτών των διαπραγματεύσεων και διαβουλεύσεων. Και όπως εδώ αναφέρθηκε και από άλλους συναδέφους εξάλλου, αποτελεί μέρος και τμήμα των στόχων της χιλιετίας που εμείς έχουμε προσυπογράψει και υποστηρίζουμε εξάλλου και έχουμε δεσμευθεί να τους προωθήσουμε, να μεριμνήσουμε και να διασφαλίσουμε την υγεία ακριβώς των γυναικών, την αναπαραγωγική υγεία όταν έρχεται η ώρα οι γυναίκες αυτές να τεκνοποιήσουν, να γεννήσουν. Πρέπει να καταπολεμήσουμε τη θνησιμότητα των βρεφών των παιδιών. Επίσης ε, και τη θνησιμότητα των γυναικών όταν πεθαίνουν την ώρα που γεννάνε παιδιά. Επίσης όσον αφορά τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία συνδέεται και συσχετίζεται και αυτή με τους στόχους αυτούς της χιλιετίας. Ευχαριστώ. Eh, σας ευχαριστούμε κυρία Πίτικεν, σας δίνω το λόγο αλλά παρακαλώ να είστε πολύ σύντομοι. Θα ήθελα να διατυπώσω μία προφορική τροπολογία. Οι συνάδελφοί μου έχουν πρόβλημα με τη λέξη provide. Αν πούμε provide δηλαδή να ισχύει ή να προσφέρει ε, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, την ε, άμβλωση, να μην πούμε provide, να πούμε support and facilitate, να στηρίξει και να διευκολύνει, πάντα αναφερόμεθα στο θέμα της άμβλωσης, αντί για provide λοιπόν, support and facilitate. Αυτή είναι η προφορική τροπολογία. So uh, Ας ψηφίσουμε λοιπόν και ευχαριστούμε την κυρία Πίτε Κέινεν. Τώρα λοιπόν ξεκινάει η ψηφοφορία, συμβαστική πρόταση παριθμών 1, παρακαλώ υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 2, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και η 6 με προφορική, προφορικές τροπολογίες. Πρώτα πρέπει να ρωτήσω κατά πόσο αν συμφωνείτε όλοι με αυτές τις προφορικές τροπολογίες. Όχι. Κάτι λέει η κυρία Λούλινγκ. Εκτός μικροφώνου δυστυχώς. Αν έχετε λοιπόν αντίρρηση, θα πρέπει να ψηφίσουμε για τις ε, προφορικές τροπολογίες. Ψηφίζουμε λοιπόν για τη συμβαστική 6. Τι έγινε τώρα. Υπάρχει αντίρρηση για την προφορική τροπολογία, οπότε δεν μπορούμε να ψηφίσουμε για προφορική τροπολογία. Πρόεδρος, σας παρακαλώ, υπάρχει αντίρρηση, άρα δεν μπορούμε να ψηφίσουμε για τις προφορικές τροπολογίες. Αυτά λέει ο κανονισμός. Ψηφίζουμε τώρα για την συμβαστική υπαριθμών 6. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 7. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα πάμε στις ε, τροπολογίες 24 λέει η πρόεδρος, μισό λεπτό. Η 33 υπέρ παρακαλώ. Η 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 34 καταπίπτει. υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 42 υπέρ κατά πρέπει να εξετάσουμε την τροπολογία υπερθμών 42 την ψηφοφορία άρχεται η ψηφοφορία ψηφίζουμε Έκλεισε. Απορρίπτεται. 10 κατά, 9 υπέρ. Η 47 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η 48 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 48 ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 11 προς 11 το αποτέλεσμα. 49 υπέρ παρακαλώ. Τα αποχές εγκρίνεται. Η 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 52 σε δύο τμήματα ψηφίζουμε. Για το πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται για το δεύτερο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 67 Πάμε στην 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 59 υπέρ κατά αποχές εγκρι... απορρίπτεται 60 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 61 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 62 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 63 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 64 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 65 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 66 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 68 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Ε, άρχεται η ψηφορία για την 68 ελέγχουμε έκλεισε η ψηφορία εγκρίνεται η 69 καταπίπτει Ε, η τροπολογία 70 υπέρ παρακαλώ κατά αποχές απορρίπτεται. Πάμε τώρα στις, στην 75 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 77 υπέρ κατά εγκρίνεται αυτή, 78 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. 79. Ψηφίζουμε για την 79 και την 89 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, η τροπολογία 95. Η ταυτόσημη, άρα μπορούμε να πάμε στην τροπολογία 85. 85 παρακαλώ. Ε, πάμε στην 85, γιατί 80 κατέπεσε, υπέρ παρακαλώ, υπέρ της 85, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Θέλετε να ελέγξουμε για την 85. Ψηφίζουμε. Ξεκινάει η ψηφορία για την 85. Ψηφίζουμε για την 87 υπέρ κατά αποχές γκρίνεται. Πάμε στην 90 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 92 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 93 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 96 και 99 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 98 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι πρέπει να ελέγξουμε ελέγχουμε για την 6 Τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και τώρα έχουμε την τροπολογία υπερτιμών 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, την 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 14 υπέρ κατά αποχές Νομίζω ότι πρέπει να ελέγξουμε. Για τη 14 ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Πάμε στην 15 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 16 καταπίπτει που σημαίνει πάμε στην 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τσεκ ελέγχουμε τη 19 Α, ψηφίζουμε τώρα έκλεισε η ψηφοφορία και απορρίπτεται η 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Υπαριθμόν 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Υπαριθμόν 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και η 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα λοιπόν έχουμε την τελική ψηφοφορία. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Έκλεισε. Και εγκρίθηκε 14 υπέρ, 6 κατά και 2 αποχές. Συγχαρητήρια ε, κύριε Κιγιόμ.